για την καταπολέμηση της παράνομης ε, μετανάστευσης. Βέβαια δεν είναι πάρα πολλοί οι Ινδοί που παράνομα βρίσκονται στις χώρες μας, αλλά υπάρχουν παρόλα αυτά, οπότε είναι θεμητό να τίθεται και αυτό σε συζήτηση. Θέλουμε επίσης να διευκολύνουμε την είσοδο φοιτητών. Γι' αυτό και αλλάζουμε κάπως το πλαίσιό μας, εφόσον αυτοί έχουν υψηλά προσόντα. Και η Ινδία θέλει να στείλει ε, φοιτητέ για έρευνα στην Ευρώπη, αλλά είναι διατεθμένη και να δεχτεί φοιτητέ από την Ευρώπη στην Ινδία. Υπάρχει η συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων και αυτό θα έπρεπε να το πλαισιώσουμε με ένα νομικό πλαίσιο που να είναι πιο αποτελεσματικό. Ευκαιρίες επίσης για τουρισμό, για επιχειρήσεις Γι' αυτό θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο περιβάλλον. Κίνα, αυτή είναι η επόμενη χώρα, με την οποία εντοπίζουμε κάποια στοιχεία προσυζήτηση προκειμένου να υπάρξει και με τη χώρα αυτή μια κοινή ημερήσια διάταξη για την μετανάστευση και την κινητικότητα με τα ίδια στοιχεία. Έχουμε κάποιες ανησυχίες με την Κίνα εξαιτία κάποιας μηνόμιμης μετανάστευσης ή επειδή υπάρχουν και κάποιες συμμορίες λαθρεμπόριου, θέλουν να διευκολυνθεί η κυκλοφορία των διπλωματών τους, οι Κινέζοι. Τα ίδια λοιπόν στοιχεία λίγο πολύ, αλλά με κάποιες μικρές διαφορές. Τρίτη χώρα μάλλον ε, για την ε, συμφωνία Ρωσία, Ουκρανία, Μολδαβία, Σερβία, Βοσνία, Μοντενέγρο, Αλβανία και Γεωργία για την διευκόλυνση θεωρήσεων. Με τις χώρες αυτές ε, συζητάμε, κυρίως με τη Μολδαβία και την Ουκρανία, αλλά και τη Ρωσία. Με την Ρωσία δεν έχουμε ολοκληρώσει τις συνομιλίες μας. Είχαμε κάποιες συνομιλίες για το περιεχόμενο της διευκόλυνσης αυτής θεωρήσεων και προτείναμε μάλιστα να αρχίσουμε και με την Λευκορωσία ε, διαπραγματεύσεις. Δεν το δέχτηκαν όμως. Οπότε σταματήσαμε. Επίσης, μόλις αυτές τις χώρες συζητούμε και το θέμα συμφωνιών ε, για τις θεωρήσεις, είτε πρόκειται για διευκολύνσεις, είτε για πανισδοχή. Οι διευκολύνσεις είναι ένα πρόγραμμα που καλύπτει τέτοια πράγματα. Μείωση του αριθμού των γράφων που απαιτούνται. Μείωση των χρημάτων που πρέπει να πληρώσει κανείς, των τελών. Να επιτρέπονται θεωρήσεις για πολλές εισόδους, για να διευκολύνονται έτσι οι επιχειρήσεις των χωρών αυτών. Το τελευταίο μου, μάλλον δύο τελευταία έχω. Το ένα είναι για την επανεισδοχή, που είναι ένα θέμα που σας έχει απασχολήσει κι εσείς. Έχουμε 13 συμφωνίες μέχρι τώρα που ισχύουν. Ο Κόγκο, Μακάο, Στριλάνκα, Δυτικά Βαλκάνια, Ρωσία, ε, Μολδοβία, Πακιστάν και Γεωργία. Έχουμε τρεις διαπραγματεύσεις δεν ισχύουν αλλά θα ολοκληρωθούν με την ε, Τουρκία για παράδειγμα και προχωράμε τις διαπραγματεύσεις με το Αζερβαϊτζάν και το Μαρόκο και αν έχουμε την συμφωνία για την κινητικότητα αυτό θα δώσει έναυσμα για να ξεκινήσουμε και αυτές τις διαπραγματεύσεις. Κάποιες από τις συμφωνίες αυτές δίνουν καλά αποτελέσματα, όπως με τη Ρωσία. Σε άλλες περιπτώσεις όμως όχι, όπως με το Πακιστάν. Γι' αυτό και πιέζουμε πολύ, προκειμένου να έχουμε αποτελέσματα. Βλέπετε, το Πακιστάν είναι μία από τις πέντε χώρες που μας ε, απασχολούν ιδιαίτερα εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τη Σρι Λάνκα, πάντως, που είχαμε μια παλιά συμφωνία που όμως δεν προχωρούσε, τις τελευταίες μέρες για πρώτη φορά έχουμε την Επιτροπή ε, Κοινής Τουρκία τώρα. Όπως γνωρίζετε έχει αρχίσει. Δεν έχει υπογραφεί η συμφωνία, αλλά έχουμε συζητήσει με τις τουρκικές αρχές. Οι διαπραγματεύσεις πάντως ολοκληρώνονται. Τέλος, διάλογος για, τις, ε, για την κατάργηση των θεωρήσεων. Έχουμε διάλογο με τη Ρωσία, την Ουκρανία, τη Μολδαβία, το Κωσυφοπαίδιο, τη Γεωργία και με την Τουρκία ελπίζω να μπορέσουμε να αρχίσουμε σύντομα. Εξαρτάται βέβαια από την υπογραφή στην Συμφωνία Επανεισδοχής. Είναι προϋπόθεση δηλαδή. Είναι προς το κοινό μας συμφέρον. Οι διαπραγματεύσεις είναι ιδιαίτερα έντονες. Για την Ουκρανία αρχίσαμε το 2008 υπήρξαν διάφορες δυσκολίες. Είναι μεγάλη χώρα. Πρέπει να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις. Το καταλαβαίνετε. Και πρόσφατα συναντιόμαστε και με τους υπουργού και βλέπουμε ότι υπάρχει πραγματική βούληση να προχωρήσουν. Μολδαβία. Προχωρήσαμε πέρυσι στο δεύτερο στάδιο και επιταχύνουμε τώρα. Υπάρχουν αποτελέσματα από τη Μολδαβία. Ανταποκρίνονται σε όλους τους στόχους. Δεν θέλω βέβαια να δώσω εγγύσει γιατί πρόκειται για μια τεχνική διαδικασία. Πιστεύουμε όμως ότι μέχρι τη διάσκεψη στο Βίλνιους για την εταιρική σχέση με τις ανατολικές χώρες θα έχει προχωρήσει αρκετά κατάσταση ώστε η Επιτροπή να μπορεί να πει ότι έχει αρκετά στοιχεία για να προχωρήσει σε πρόταση. Κωσυφοπαίδιο. Ήμουνα στο Κωσυφοπαίδιο πριν από μερικές εβδομάδες. Υπάρχει ένα ειδικό πρόγραμμα σε ένα δύσκολο πλαίσιο. Είχαμε 70 συστάσεις που έχουν να κάνουν με τους θεσμούς και την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Η συμμετοχή όμως είναι πολύ καλή από την άλλη πλευρά. Και οι αρχές της χώρας δείχνουν ότι το θέλουν πολύ. Η Γεωργία. Χθε στο Συμβούλιο συζητήσαμε. Η Επιτροπή θα δώσει το πρόγραμμα δράσης τη Δευτέρα για την ε, διευκόλυνση θεωρήσεων. Και έτσι και αυτή η διαδικασία θα έχει καταλήξει. Ελπίζουμε γρήγορα. Εδώ ολοκληρώνω. Θα μπορούσα να σας δώσω πολλές λεπτομέρειες ακόμα, αλλά καλύτερα να απαντήσω σε ό,τι ερωτήσεις έχετε, εφόσον θέλετε. Ελπίζω και την επόμενη φορά θα ξεκινήσουμε με την Τουρκία. Πάντα λέμε ότι είναι μια σημαντική στιγμή. Είναι σημαντικός εταίρος και στα πλαίσια της Σας Ευχαριστώ. Uh, ευχαριστώ πολύ. Θα πάμε αμέσως στις ε, ομιλίες των εισηγητών. Η κυρία Ζόμερ είναι πρώτη. Για συμφωνία Ευρωπαϊκής Ενώσεως και Δημοκρατία της Τουρκίας για την επανειστοχή ατόμων που διαμένουν άνευ αδεία. Κυρία Ζόμερ, έχετε το λόγο. Yeah, uh, Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η συμφωνία επανειστοχής με την Τουρκία Ήταν μια μακρά ιστορία, Οχτώ χρόνια διαπραγματεύσαμε την Τουρκία, ένας πολύ μεγάλος χρονικός ορίζοντας. Πέρσι κλείσαν οι διαπραγματεύσεις για το θέμα αυτό. Αλλά έκτοτε, για να το διατυπώσω επιφυλακτικά, φαίνεται ότι η Τουρκία δεν είναι έτοιμη να υπογράψει τη συμφωνία αυτή. Η Τουρκία εξαρτά την υπογραφή αυτής της συμφωνίας από διευκολύνσεις προξενικών θεωρήσεων και απαλλαγή από προξενικές θεωρήσεις. Το πρόβλημα λοιπόν που αντιμετωπίζουμε είναι ότι δεν είναι όλα τα κράτη-μέλη έτοιμα να δεχτούν ότι θα πρέπει να συμφωνήσουν σε αυτήν την φιλελευθερωποίηση για τις προξενικές θεωρήσεις για τους πολίτες της Τουρκίας. Και επομένως <clears throat> είναι εν αμφισβητήσει σοβαρά το θέμα της συμφωνίας επανεισδοχής. Εμείς γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή ότι είναι πολύ μεγάλη η παράνομη ε, μετανάστευση στην Ευρώπη που προέρχεται από τα χερσαία σύνορα της Τουρκίας με την Ελλάδα και τα θαλάσσια σύνορα φυσικά και ε, υπάρχει και η, εντύπωση και η υποψία σε πολλούς ότι οι Τούρκοι αφήνουν τα σύνορα να είναι ιδιαίτερα διαπερατά λόγω της προσπάθειάς τους να εξασφαλίσουν την φιλελευθερωποίηση στον τομέα των προξενικών θεωρήσεων. Αυτό αποτελεί μια μορφή εκβιασμού βέβαια, το έχω πει και στην τουρκική πλευρά. Εν πάση περιπτώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τίθεται υπό πίεση γιατί εμεί φυσικά χρειάζεται να εξασφαλίσουμε την εφαρμογή αυτής της συμφωνίας. Όλα αυτά είναι εντυπωσιακά βέβαια γιατί η Τουρκία είναι μια, μια χώρα υποψήφια για την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την άλλη πλευρά, για τους Τούρκους δεν είναι ιδιαίτερα σαφές το γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαπραγματευτεί συμφωνίες για διευκόλυνση προξενικό θεωρήσεων με όλες τις άλλες υποψήφιες χώρες, αλλά για την Τουρκία έχει ειδικέ απαιτήσει. Εγώ Φαίνω, θα ήθελα να έχω και την άποψη του εκπροσώπου τη Κομισιόν, γιατί αυτή τη στιγμή φαίνεται λόγω των διαφορετικών απόψεων των κρατών μελών να μην είναι ανοιχτό ο δρόμο για μια συμφωνία, για την εφαρμογή τη συμφωνία επανεισδοχή. θα με ενδιαφέρει επίση να γνωρίζω ποιε είναι οι θέσει στο Συμβούλιο Υπουργών για τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ. Την κυρία Μπάουρ θα καλέσω τώρα που είναι και για τη διευκόλυνση των θεωρήσεων με την Αρμενία και την ε, Συμφωνία Επανεισδοχής με την ίδια χώρα. Η κυρία Μπάουρ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για τις πληρέστατες εξηγήσει για την ε, όλη κατάσταση. Μας είπατε ότι με τη Ρωσία τα πράγματα πηγαίνουν καλά όσον αφορά την επανειστοχή. Με το Πακιστάν πάνε άσχημα τα πράγματα. Με την Αρμενία τι γίνεται. Στο έγγραφό μας αναφέρει ότι οι τελευταίες διαπραγματεύσεις έλαβαν χώρα στις 12 Οκτωβρίου. Ποια είναι η κατάσταση τώρα. Έχουμε το θέμα της διευκολύνσεως των θεωρήσεων με προθεσμίες για σύνταξη εκθέσεως την 5 Μαρτίου χωρίς συμφωνία επανεισδοχής αυτό είναι αδύνατον. Αδύνατο να προχωρήσουμε. Η ερώτησή μου είναι ποια είναι η κατάσταση σε αυτό το ζήτημα. Και άλλο ερώτημα. Φαίνεται να είναι τεχνικής φύσεως, αλλά κατά κάποιο τρόπο είναι ενδιαφέρουσα. Και περιμένω να ακούσω τις εξηγήσεις σας. Στη Συμφωνία Διευκολύνσεως Θεωρήσεων χρησιμοποιείται κάποια διατύπωση που αφορά την ηθαγένεια. Αναφέρεται τους πολίτες. Στη Συμφωνία Επανιστόχης χρησιμοποιείται συνεχώς η υπηκότητα. και σε μία σειρά, σε μία παράγραφο βάζεται ηθαγένεια και σε άλλη υπηκότητα. Για ποιο λόγο φαίνεται να είναι ισότιμη η όρη. Γιατί υπάρχει διαφοροποίηση. Στο ένα έγγραφο λέτε citizenship και στο άλλο έγγραφο λέτε nationality. Υπηκότητα και ηθαγένεια. Είναι τεχνικής φύσεως το ερώτημα. Ενδιαφέρον ζήτημα. Το βασικό ερώτημα για την ώρα είναι μπορούμε να προχωρήσουμε με αυτό το ζήτημα ή όχι. Ποια είναι η κατάσταση αυτό το ερώτημα. Ευχαριστώ πολύ. Όσον αφορά, αν συμφωνεί ο κύριος Μαρινέσκου, θα ήθελα να τον καλέσω σαν τρίτο εισηγητή. Η διαφορά είναι ότι έχετε ήδη κάποιο κείμενο, ενώ εμείς απευθύνουμε ερωτήσεις προς την Επιτροπή. Θα σας ζητήσω να κάνετε τώρα την παρουσίαση, ούτω ώστε να έχουμε μια σφαιρική εικόνα για τη συζήτηση. Δεν ναι, μπορώ να το κάνω, λέει ο Μαρινέσκου. Μου ζητήθηκε πράγματα ετοιμάσω ένα κείμενο, να το στείλω, μου το ζήτησε η Γραμματεία. Ευχαριστώ πολύ για την ε, παρουσίασή σας. Συμφωνώ ότι η, Μολδαβία, η Μόλδοβα μάλλον ε, κάνει αυτά που πρέπει ε, και ελπίζω να ολοκληρωθεί η συμφωνία μέχρι τη συνεδρίαση στο Βίλνιους, όχι μόνο από τεχνική σκοπιά, αλλά στο σύνολό της. Έχουμε σύσταση του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, από το Φεβρουάριο να γίνει αυτό. Όσον αφορά την απόφαση του Συμβουλίου για τη διευκόλυνση των θεωρήσεων, νομίζω ότι είναι πολύ καλή απόφαση, οπότε οι Μολδαβοί πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν άνευ θεωρήσεως, αν κατέχουν βιομετρικό διαβατήριο. και για την χορήγηση θεωρήσεων μειώνονται οι προδιαγραφές. Δεν πρέπει να πηγαίνουν αυτοπροσώπως στο γραφείο για να παραλάβουν τη θεώρηση και μπορούν να μπορεί να υποβληθεί το αίτημα από ε, Μολδαβούς που είναι και Ευρωπαίοι πολίτες και Μολδαβούς που ε, διαμένουν αλλού. Ισότιμη είναι η αντιμετώπιση τώρα όσον αφορά τους Ρώσους και τους Μολδαβούς, διότι αυτό ε, αποτελούσε πρόβλημα. Κυρίως για τους Μολδαβούς πολίτες που θέλαν ρωσικό διαβατήριο μόνο και μόνο για να έχουν ευκολότερη πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι το μόνο σχόλιο που έχω. Ε, ελπίζω να καταβάλλετε κάθε προσπάθεια για να συναυτεί αυτή η συμφωνία με τη Μοδαβία στο... μέχρι να πραγματοποιηθεί το φθινόπωρο η συνάντηση αυτή στο Βίλνιος. Ευχαριστώ. Ίσως θα ήταν χρήσιμο. Πρωτού ξεκινήσουμε τη συζήτηση ο κύριος ε, Ματσερβίτσι να απαντήσει εν συντομία τα ερωτήματα τα οποία έχουν απευθυνθεί προς αυτόν και αυτή τη στιγμή έχω μονάχα μία αίτηση για λήψη του λόγου από τους συναδέλφους. Σηκώστε την κάρτα σας αν θέλετε να λάβετε το λόγο. Κύριος Ματσερβίση πρώτα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ξεκινώ με τα ερωτήματα με τη σειρά που διατυπώθηκαν. Πρώτα η Τουρκία. Είναι δύσκολη η σχέση μας με την Τουρκία. Είναι μια πολύπλοκη χώρα και πολύ καλοί διαπραγματευτές και φυσικά εμπλέκονται πάρα πολλά στις διαπραγματεύσεις. Ε, <clears throat> υπάρχει μεγάλος βαθμός ολοκλήρωσης που έχει επιτευχθεί σε οικονομικό επίπεδο, αλλά είναι μια πολύπλοκη σχέση που έχουμε με την Τουρκία. Το γεγονός είναι ότι η συμφωνία επανεισδοχής έχει μονογραφηθεί. Υπάρχει το τελικό κείμενο δηλαδή. Και εγώ το μονογράφησα ως ε, ως κύριος διαπραγματευτής και από τον Τούρκο πρεσβευτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχει κανείς λοιπόν ο οποίος διαφυσβητεί το κείμενο. Το κείμενο αυτό όμως πρέπει κάποια στιγμή να, να υπογραφεί και μετά να εφαρμοστεί. Το ερώτημα είναι πώς αυτή η συζήτηση μπορεί να συνδυθεί με αυτά που έχουμε αναφέρει για, την, για τον ορίζοντα, την προοπτική της πλήρης φιλελευθερωποίησης για τις προξενικές θεωρήσεις, όχι μόνο χατή διευκόνηση γιατί οι ενδιάμεσες λύσεις δεν θεωρούνται από την τουρκική πλευρά επαρχής και ενδιαφέρουσες. Οι δύο ενέργειες λοιπόν θα πρέπει να γίνουν ταυτόχρονα. Όταν ξεκινήσουμε το διάλογο για τη φιλελευθερωποίηση των προξενικών θεωρήσεων, τότε συγχρόνως η Τουρκία θα πρέπει να υπογράψει και να θέσει σε εφαρμογή τη Συμφωνία Επανεισδοχής. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι υπό αμφισβήτηση. Επομένως, αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι να διευκρινίσουμε ορισμένα σημεία τα οποία θα ζητήσουμε από την Τουρκία να κάνει μέσα στα πλαίσια του κανονικού διαλόγου για τη φιλελευθερωποίηση των προξενικών θεωρήσεων τα θέματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια εγγράφων κτλ. Πρέπει όμως οι δύο διαδικασίες να προχωρήσουν παράλληλα. Η δική μου πρόβλεψη είναι ότι, και αυτά είναι πολύ καλά κατανοητά από την τουρκική πλευρά, δεν υπάρχει κάποια ιδέα να δημιουργήσει η Τουρκία μια ασυμμετρία στην εφαρμογή αυτών των μέτρων. Αυτό το οποίο συζητούμε σήμερα είναι τι προβλέπεται να ζητήσουμε από την Τουρκία για να συμμορφωθεί με τις βασικές προϋποθέσεις με, για την ε, φιλελευθέρωση προξενικών θεωρήσεων σε ένα επίπεδο το οποίο είναι ε, προσιτό για αυτούς σε οικονομικό επίπεδο. Θα πρέπει να προχωρήσουν και οι δύο διαδικασίες από κοινού και επομένω, είμαστε απόλυτα σε συμφωνία με αυτά που έχουν αποφασιστεί από το Συμβούλιο και από την Τουρκία. Είναι σαφής οι κανόνες του παιχνιδιού. Το θέμα είναι πότε μπορούμε να ξεκινήσουμε το παιχνίδι αυτό. Το παιχνίδι μπορεί να λειτουργήσει μόνο αν, ξε, αν μπορούν να ξεκινήσουν και δύο διαδικασίες εν παραλίδο. Αυτό που κάνει τώρα η Τουρκία σε σχέση με τον αγώνα κατά της παράνομης μετανάστευσης και τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάνει πολλά πράγματα η Τουρκία. Πρώτα απ' όλα ξέρετε ότι η Τουρκία κάνει τεράστια προσπάθεια για να υποδεχθεί τους πρόσφυγες από τη Σύρια. Και αυτό είναι κομμάτι του παιχνιδιού. Γιατί πολλά από τα κράτη-μέλη μας θα υφίστανται πάρα πολύ ισχυρή πίεση για να υποδεχθούν όλους αυτούς τους πρόσφυγες. Τα κάνει αυτά η Τουρκία με τα πιο υψηλά πρότυπα. Αυτό λοιπόν πρέπει να αντιμετωπιστεί σαν τμήμα της συνολικής εικόνας, ακόμα και αν είναι ένα παράπλευρο θέμα. Γιατί αργά ή γρήγορα θα πρέπει να δούμε πώς θα εφαρμόσουμε την αρχή της προστασίας για τα άτομα αυτά. Η Τουρκία κάνει λοιπόν πάρα πολλά πράγματα ήδη. Ένα δεύτερο σημείο. Υπάρχει καλή συνεργασία στη διαχείριση των συνόρων και την ε, τον αγώνα κατά της παράνομης μετανάστευσης. Υπάρχει ένα μνημόνιο αναγνώρισης μετα... μεταξύ τη Frontex και της Τουρκία και μια αποστολή της Frontex θα πάει την επόμενη εβδομάδα στην Τουρκία για να προωθήσει τα θέματα αυτά. Υπάρχει μια κόκκινη γραμμή μεταξύ των δύο πλευρών που είναι πάντα ανοιχτή. Προχωρούν τα πράγματα. Η συμφωνία <clears throat> επανεισδοχής υπάρχει αυτή τη στιγμή σε επίπεδο διμέρε μεταξύ πολλών χωρών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, παραδείγματο χάρη Ελλάδο και Τουρκία, λειτουργεί. Όχι πάντα με άψογο τρόπο, με πλήρη σεβασμό των κανόνων, αλλά αυτό είναι τμήμα τη συζήτηση που κάνουμε τώρα και η τουρκική πλευρά αντιμετωπίζουν με ανοιχτό πνεύμα. Είναι πολύ καλή συνεργασία επίση <clears throat> και η συνεργασία για την σύλληψη των παρανόμων μεταναστών που προσπαθούν να φτάσουν στα θαλάσσια ή στα χερσαία σύνορα της Τουρκίας. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι απαραίτητη η συμφωνία επανιστοχής για να έχουμε και μια επιτροπή επανεισδοχής που να μπορεί να συζητήσει τα έκρεμή προβλήματα. Υπάρχουν πολιτικά προβλήματα, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει και κάποια πρόοδος. Επομένως εγώ είμαι αν σίγουρα ήμουν έτοιμος να περατώσω τη διαδικασία αυτή επανεισδοχής σε τεχνικό επίπεδο να προετοιμάσω και ένα εθνικό σχέδιο το, για την Τουρκία το οποίο ενεκρίθηκε από το Συμβούλιο. Μετά από όλα αυτά, επιτρέψτε μου να είμαι αισιοδόξο και για το μέλλον. Για την Αρμενία. Αν λειτουργεί η Συμφωνία Περιστοχή, λειτουργεί. Χίλια δέκα άτομα επανεπατρίστησαν στην Αρμενία πέρσι βάσει αυτού του, αυτής της συμφωνίας και Υπάρχουν περίπου 2.000 άτομα τα οποία συνελήφθησαν ως ε, παράνομοι μετανάστες. Υπάρχει πάντα ένα χάσμα βέβαια μεταξύ αυτών οι οποίοι συλλαμβάνονται και αυτοί, αυτών οι οποίοι επιστρέφονται. Για τη διαφορά μεταξύ υπηκότητος και εθνικότητος. Για μας δεν υπάρχει καμία διαφορά. Χρησιμοποιούμε ίσως διαφορετικές εκφράσεις τις φορές, αλλά υπάρχει, δεν υπάρχει καμία διαφορά. Για τη Μολδαβία, <clears throat> όταν λέω ότι στο Βίλνιος θα μπορέσουμε να κλείσουμε τουλάχιστον τις τεχνικές πτυχές. Το λέω γιατί δεν είναι μονάχα μία διαπραγμάτευση. Αυτό που λέμε διαπραγματεύσεις είναι μονάχα προπαρασκευαστικές ενέργειες για να μπορέσει η Κομισιό να κάνει μια πρόταση προς το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε μια εσωτερική διαδικασία και ιδίω να περάσει αυτή η διαδικασία από του συνομοθέτε, από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Μέχρι τότε δεν είναι δυνατόν να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Μπορούμε να πούμε ότι έχουμε κλείσει τι διαπραγματεύσει με την έννοια του ότι οι επαφέ μα μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Μολδαβία είχαν σαν αποτέλεσμα να μπορούμε να πούμε την επόμενη εβδομάδα ότι μπορεί η Κομισιό να υποβάλει μια πρόταση στο Συμβουλίο και το Κοινοβούλιο. Αλλά δεν μπορώ να προχωρήσω περισσότερο. Κατά τα άλλα, υπάρχει καλή αμοιβαία κατανόηση. Είναι πολύ σημαντικέ οι μεταρρυθμίσει που έχουν γίνει. Αν συνεχίσουμε λοιπόν αυτό το ρυθμό, πιστεύω ότι μέχρι την ε, ανάληψη πριν από τη συνάντηση του Βίλνιους θα έχουν λυθεί όλα αυτά τα πράγματα. Ευχαριστώ. Έξι έχουν ζητήσει το λόγο. Επτά. Συμπεριλαμβανομένη κυρία Ζόμερ. Θα ακούσουμε πρώτα τους άλλους, αν συμφωνείτε, και στο τέλος ε, παίρνετε το λόγο. Η κυρία Λόπες, ο Μέρο Λόπες έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Μανσερβίση, για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Δύο θέματα θέλω να σας ρωτήσω. Πρώτον, για τη συμφωνία με το Μαρόκο. Μπορείτε να μας πείτε ποια είναι τα πιο δύσκολα, τα πιο επίμαχα σημεία για να καταλήξουμε σε συμφωνία για την κινητικότητα. Καταλαβαίνετε, επειδή είναι τόσο κοντά στην Ευρώπη, μας ενδιαφέρει. Επίσης, επειδή έχει ως χαρακτηριστικό η χώρα αυτή να έχει πάντα ανοιχτά σύνορα και με το Μαλί, τον πόλεμο εκεί, με την τρομοκρατία στο Σαχέλ, υποθέτω ότι θα υπάρχει πρόβλημα προσφύγων. Πώς το λαμβάνετε αυτό υπόψη σας στη συμφωνία που διαπραγματεύεστε. Δεύτερον, Τουρκία. Γιατί για να, να μπει κανείς στην ε, Τουρκία δεν χρειάζεται τίποτα, 30 ευρώ. Δηλαδή οποιοδήποτε μπορεί να αγοράσει την θεώρηση που απαιτείται και να μπει στην Τουρκία. Ε, πώς γίνεται. Υπάρχουν πολλοί πολίτες από πάρα πολλές ε, χώρες που δεν έχουν πόλεμο, γιατί βέβαια ορισμένοι έχουν ε, έτσι, Συρία, Αφγανιστάν κτλ. Ενώ άλλοι, Δουμενικανική Δημοκρατία, Αλγερία. Και τελικά καταλήγουν στην Ελλάδα όλοι αυτοί. Στην Τουρκία δεν έχουν κανένα πρόβλημα να μπουν. Μπαίνουν πολύ εύκολα. πώς είναι δυνατόν ε, να μιλένε ότι περνάνε από την Τουρκία όλοι αυτοί που καταλήγουν τελικά στην Ελλάδα. Τι ε, προϋποθέσεις πάνω, τι προδιαγραφές βάζετε εσείς για την επανιστοχή. Ελλάδα, Μάλτα, όλες οι χώρες ε, του Νότου υποφέρουν πάρα πολύ από αυτήν την παράνομη μετανάστευση. Εμείς μιλάμε για τη μετανάστευση και την κινητικότητα, αλλά 15 χρόνια τώρα το θέμα των προσφύγων δεν έχει, δεν το έχουμε χειριστεί και η διεθνής προστασία πώς θα την προσφέρουμε. Υπογράφουμε τη μία συμφωνία μετά την άλλη. Έχουμε δεκάδες χιλιάδες τα διάφορα κέντρα για τους πρόσφυγες που τελικά ε, τους κρατάμε φυλακισμένους ακόμα και δεν είναι εγκληματίες. Και όταν μιλάμε λοιπόν για τη μετανάστευση και την κινητικότητα, πρέπει να μιλάμε και για τους πρόσφυγες. Εντάξει, η Frontex προσπαθεί εδώ και μερικά χρόνια, συνεργάζεται με τις αρχές των χωρών αυτών, αλλά οι χώρες του Νότου, δεν έχουν καταφέρει να αποφεληθούν αρκετά έχουν πολύ χαμηλή βοήθεια σε σχέση με τις παραδοσιακές χώρες όπως είναι η Ολλανδία, η Αγγλία κτλ. Πολύ λιγότεροι θέλουν να πάνε εκεί, αλλά εκεί καταλήγουν. Πάνω σε αυτό πρέπει να δουλέψουμε λοιπόν. Γιατί δεν συνεργαζόμαστε περισσότερο με τις χώρες του Νότου. Δεν είναι μόνο θέμα αλληλεγγύης, είναι ότι τελικά ε, το καθεστώς του πρόσφυγα για να το δώσει μια χώρα πρέπει να έχει δυνατότητα να τους απορροφήσει. Η υπηρεσία ασύλου δεν έχει προπολογισμό, ενώ η Frontex έχει. Η υπηρεσία ασύλου δεν έχει. Ήρθε εδώ και μας μίλησε ο υπεύθυνο, μας είπε πόσο λίγοι είναι. Πώς θα χειριστούμε λοιπόν το θέμα της διεθνούς προστασίας όταν δεν υπάρχουν χρήματα, αν δεν υπάρχει προσωπικό. Και στην Ελλάδα δεν έχουν τίποτα από όλα αυτά είναι τραγική κατάσταση. Πήγαμε, ταξιδέψαμε και την είδαμε την κατάσταση. Δεν, δεν είμαστε καθόλου αισιόδοξοι. Κύριε Μανσερβίση, αν η Ευρώπη δεν ε, βοηθήσει, οι μεγάλες δηλώσεις είναι περιτές. Χρήματα χρειάζονται. Χρήματα και συγκεκριμένη βοήθεια προς αυτές τις χώρες. Ευχαριστώ κυρία Ντάνοκα είναι η επόμενη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και μας Σερβίση για την παρουσίαση. Έχω μία λεπτό συγκεκριμένη ερώτηση και μία γενικότερη για την Αρμενία πρώτα απ' όλα και την επανεισδοχή. Έχετε στοιχεία σχετικά με προβλήματα επανεισδοχής ανθρώπων από τον Αγκόρνο Καραμπάχ. Φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν προβλήματα όπως ε, όταν συζητούσαμε για την επανειστοχή στη Γεωργία. Από, για αυτούς που έρχονται από την Αυχασία, παραδείγματος χάρη. Είναι θέμα έλλειψης ταξιδιωτικών εγγράφων, τόπο κατοικίας, ε, υπηκότητα, ίσως οδηγεί αυτό σε προβλήματα σε κάποιον που πρέπει να επιστρέψει στο Αζερμπαϊτζάν, στην Αρμενία κλπ. Είναι ένα πρόβλημα αυτό που συζητάτε ή όχι. Δεύτερον ερώτημα. Έχουμε έξι, έξι χώρες ε, ε, ε εταιρικής σχέσης με τις χώρες και τη Ρωσία. μπορεί να συγκρίνεται αυτές τις χώρες όσον αφορά τη συμφωνία για την ελάφρυνση απαιτήσεων για τις θεωρήσεις. Εμείς θα θέλαμε να εναρμονιστούν οι συμφωνίες. Αυτή θα έπρεπε να είναι η πολιτική μας. Το κάνουμε αυτό. Ευχαριστώ. Η κυρία Κέλλερ έχει το λόγο. Thank you. Ευχαριστώ μόνο ένα ερώτημα, το οποίο είναι πολύ συγκεκριμένο. Πριν από ένα χρόνο και παραπάνω συζητήσαμε την ε, αξιολόγηση των συμφωνιών επανιστοχής. Η Κομισιόν έκανε μια αξιολόγηση όπου περιλάμβανε ορισμένε προτάσεις για το τι θα έπρεπε να αλλάξει. Φαίνεται ότι κανείς δεν είχε χρησιμοποιήσει τα κρατημέλη τη ρήτρα υπηκόου τρίτης χώρας. Και προβλεπόταν να μην ξαναμπεί αυτό στις συμφωνίες επανιστοχής και ορισμένες άλλες προτάσεις. Τι έχει γίνει με όλα αυτά. Τι έγινε με αυτές τις προτάσεις θα υπάρξει μια μεταρρύθμιση στη Συμφωνία επανεισδοχής. Τα διδάγματα αυτά έχουν ενσωματωθεί σε αυτές που διαπραγματεύεστε τώρα, που σχεδιάζετε να διαπραγματευτείτε. Κυρία Ένστ. Ευχαριστώ. Η συμφωνία περιστοχής με την Τουρκία είναι ένα πολύ μεγάλο εγχείρημα εναντί των αντίστοιχων συμφωνιών με άλλες χώρες και έχει πολλές επιπτώσεις και σε ανθρώπινο επίπεδο. Και επομένως, όπως έρχομαι στο εξή θέμα, ναι, λέτε ότι η Τουρκία ζητά την ε, φιλελευθερωποίηση στις ε, προξενικές θεωρήσεις, το καταλαβαίνω αυτό. Ποιες άλλες πτυχές έχουν παίξει ρόλο σε αυτές τις διαπραγματεύσεις με την Τουρκία. Τι θα προκύψει λοιπόν όταν γίνει αυτή η συμφωνία για την επαρισδοχή. Ο κ. Παπα-Νικολάου. Once more, thank you, Mr. Ευχαριστώ πάλι κύριε Μαντσεβίτσι για την παρουσίασή σας, για την σας αυτές. Θα μιλήσω για την Τουρκία. Είπατε ότι παίζετε ένα παιχνίδι με δύο παίκτες. Αναρωτιέμαι αν αυτό το παιχνίδι παίζεται με δίκαιους, με τίμιους κανόνες. Η τελευταία συμφωνία που είχαμε, όπως αναφέρεται στο κείμενο, υπάρχει μία ρήτρα ότι θα πρέπει να υπάρξει μια τριετής μεταβατική περίοδος για την Τουρκία, ώστε η Τουρκία να μπορέσει να δέχεται υπηκόους τρίτων χωρών στο έδαφος της, όταν <clears throat> έχουν έλθει στην Ευρώπη παράνομα. Χρειαζόμαστε τουλάχιστον δύο χρόνια για να, τελειώσει η διαπραγμάτευση και η, και η εφαρμογή αυτής της συμφωνίας και άλλα τρία χρόνια για να πάρει πίσω η Τουρκία τους υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν έρθει παράνομα στην Ευρώπη. Ας πούμε ότι προσπαθούμε να πετύχουμε αυτή τη διαπραγμάτευση επειδή δεν έχουμε άλλη επιλογή. Πώς είναι αυτό ένα δίκαιο παιχνίδι όταν η Τουρκία θέλει από την πρώτη μέρα που θα εφαρμοστεί η συμφωνία να έχει μια φιλελευθερωποίηση ε, των προξενικών θεωρήσεων όταν οι παράνομοι μετανάστες που έρχονται από την Τουρκία είναι πάνω από το 90%. Δηλαδή ουσιαστικά αφήνουμε το 90% εκρεμές στον αέρα για 5 χρόνια και έχουμε μια ρύθμιση μόνο για το 10% και από την άλλη μέρα έχουμε μια φιλελευθερωποίηση σε επίπεδο προξενικών θεωρήσεων. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση, αλλά με έναν τρόπο ο οποίος θα είναι πιο δίκαιος. Ας αφήσουμε λοιπόν εκρεμεί τη διαδικασία φιλελευθεροποίησης για τις υποξερικές θεωρήσεις για κάποιο διάστημα, αν θέλουμε το παιχνίδι να είναι ισοδίκαιο. Θα ήθελα να ξέρω και την άποψή σας και για το εξή. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή είναι σε μια διαδικασία που θα πάψει να ζητά προξενικές θεωρήσεις με γειτονικέ της χώρες έχουν κάνει συμφωνία με την, ε, με την Νότια Αφρική για να έρχονται χωρίς βίζα οι πολίτες αυτών χωρών και τώρα είναι υποδιαπραγμάτευση συμφωνίες με το Ιράκ και το Ιράν. Θα περνάνε στην Τουρκία λοιπόν όλοι αυτοί οι άνθρωποι και κάποια στιγμή μετά θα περνάνε σε εμά. Σίγουρα κάνει πολλά πράγματα η Τουρκία για τη Συρία και τους πρόσφυγες και μπορώ να το σεβαστώ αυτό. Επίσης υπάρχει βελτίωση στη συνεργασία των ε, τουρκικών αρχών για τη φύλαξη των συνόρων. Ένα τελικό σχόλιο. Ξέρουμε ότι η Ευρώπη υποστηρίζει την Τουρκία στην διαδικασία εξασφάλισης των συνόρων ως υποψήφια χώρα και μπορεί να υποφελθεί και από την χρηματοδότηση που έχει ως υποψήφια χώρα. Όταν πήγαμε στον Εύρο, δεν θυμάμαι αν ήταν παρόντες, αν το θυμούνται οι άλλοι συνάδελφοι που ήταν που είναι παρόντες εδώ. Όταν είδαμε τον ε, φράχτη ο οποίος έχει δημιουργηθεί στη βόρεια μεθοριακή περιοχή, εμφανίστηκαν στρατιωτικά οχήματα του τουρκικού στρατού μας παρακολουθούσαν καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Γιατί δεν γίνεται αυτό όταν έρχονται οι λαθρέμποροι με τους παράνομους μετανάστες. Έχουμε κάποιες πληροφορίες για την Τουρκία σε σχέση με τους λαθρεμπόρους ανθρώπων. Πώς μπορεί κανείς να ξεκινήσει από την, βόρεια, από νότια Τουρκία να φτάσει μέχρι τη βόρεια Τουρκία χωρίς να αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Εγώ σέβομαι τις προσπάθειες που καταβάλει η Τουρκία σε αυτή τη χρονική εποχή Υπάρχει ε, βελτίωση, αλλά αυτό δεν επαρκεί αυτή τη στιγμή και δεν αποτελεί πρόσχημα. Ζητώ συγγνώμη από την κυρία Γκρίσμπεκ. Ε, ε, σας, δεν σας είδα πριν, σας έχω επόμενη στον κατάλογο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε για τις εξηγήσεις που μας δώσατε και για τη σφαιρική παρουσίαση των διαπραγματεύσεων ε, για τη συμφωνίες. Σαν η συγγήτρια, σκιώδη συγγήτρια για την επανειστηχή για τη συμφωνία με την Τουρκία. Μετά τις πρώτες παρατηρήσεις δώσατε κάποιες απαντήσεις στα ερωτήματα που μου είχαν δημιουργηθεί. Όσον με αφορά, θα ήθελα να γνωρίζω το μηχανισμό συμμετρίας μεταξύ απελευθέρωσης των καθεστώτων των θεωρήσεων και των συμφωνιών επανεισδοχή. Απαντήσατε με μεγάλη σαφήνεια εξηγώντα ότι δεν υπήρχε ασυμμετρία, ότι ακόμα και αν οι συνθήκε και των διαπραγματεύσεων ήταν περίπλοκες και δύσκολε, αυτό ισχύει με όλου του εταίρου πιστεύω, παρόλα αυτά τα πράγματα προχωρούσαν είπατε. Εξετίμησα το ότι υπογραμμίσατε την απάντηση που έδωσε η τουρκική κυβέρνηση όσον αφορά τις δεκάδες χιλιάδες ε, Συρίους ε, που είναι στα σύνορα μεταξύ Τουρκίας και Συρίας και που επιτρέπει σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους να ζήσουν έναντι της αδράνειας της διεθνούς ε, κοινότητας. Σας ευχαριστώ για τη σαφήνεια των όσων μας είπατε. Δράτω με τις ευκαιρίες, παρόλο που το παιχνίδι συνίσταται στο να υποβάλλουμε ερωτήσεις, θα ήθελα όσον αφορά αυτό που αναφέρατε για τις διαπραγματεύσεις με το Πακιστάν. Το 2010 στη συζήτηση για τη Συμφωνία Επανεισδοχής με το Πακιστάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε έναντι του Κοινοβουλίου. Θα θυμόσαστε ότι υπήρξαν πολλά ερωτηματικά τότε και μεγάλη αντίσταση όσον αφορά αυτή τη συμφωνία που ήταν ε, κάτι σαν εκρηκτικό θέμα και δεσμεύτηκε έναντι του Κοινοβουλίου ε, να δώσει πληροφορίες, λεπτομερείς πληροφορίες, επίκαιρες, εμπεριστατωμένες όσον αφορά την εφαρμογή των συμφωνιών επανεισδοχής. Και όχι μόνο ε, την πορεία των διαπραγματεύσεων, αλλά περισσότερο να αφορούν οι πληροφορίες στην συγκεκριμένη εφαρμογή με αριθμητικά στοιχεία ή δυνατόν. Πρακτική εφαρμογή των διαφόρων συμφωνιών και νομίζω ότι είναι σημαντικό για όλους τους ε, συναδέλφους αυτό για να μπορέσουν να τοποθετήσουν τοποθετούνται σωστά, να έχουν τις πληροφορίες, να μπορούν να τοποθετούνται έχοντας επίγνωση των γεγονότων για τις συμφωνίες. Προσωπικά ανησυχώ κάπως λόγω της ελλείψης πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση που αφορά την προστασία των ανθρώπων που έτυχαν επανεισδοχής στο Πακιστάν. Η Επίτροπος, η κυρία Μέλστρομ, ανέφερε αυτό που είπατε κι εσείς. Το αναφέρατε τότε και το αναφέρατε εκ νέου τον Ιούλιο 2012, αν δεν σφάλω, όταν περιγράψατε κάτι τελευταία ενημέρωση, ίσως να κάνω την ημερομηνία, τέλο πάντων τότε μας μιλήσατε για ένα πιλωτικό σχέδιο ε, στο Πακιστάν για να υλοποιούνται οι αποφάσεις που λαμβάνουμε εδώ και να δούμε ποιε συγκεκριμένε ε, συνέπειε που έχουν σαν αφορά του ανθρώπους. Και ο, το Πακιστάν είναι ένα από τα πολλά παραδείγματα ε, που έχουμε, που υπάρχουν άνθρωποι εκεί που είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Θα θέλαμε λεπτομερά αριθμητικά στοιχεία τι γίνεται με τα άτομα που, ε, που επιστρέφουν στο Πακιστάν, που γίνεται επανιστοχή στο Πακιστάν και είναι προαπαιτούμενο αυτό για να μπορώ να τοποθετήσω κι εγώ. Ευχαριστώ και στο τέλος η κυρία Ζόμερ θέλει να ξαναμιλήσει. Ja, Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να σας ευχαριστήσω και για τα ερωτήματα για μας ελβήσει. Ένα ερώτημα δεν το απαντήσατε όμως κατά την εντύπωσή μου. Ποια είναι η κατάσταση στο Συμβούλιο σε σχέση με τη φιλελευθερωποίηση των προξενικών θεωρήσεων για την Τουρκία. Γιατί είναι απόλυτα σαφές ότι η Τουρκία δεν θα δεχτεί τη Συμφωνία Επανεισδοχής χωρίς τη φιλελευθερωποίηση. Αυτή είναι η θέση της Τουρκίας. Εσείς τώρα βλέπετε στο Συμβούλιο κάποια δυνατότητα να υπάρξει μια συμφωνία για το θέμα αυτό. Ξέρουμε όλοι ότι είναι πολύ το ζήτημα αυτό. Αλλά ξέρουμε ότι υπάρχουν ανησυχίες στα κράτη-μέλη για το θέμα αυτό και ιδίως σε ορισμένα κράτη-μέλη όπου υπάρχουν ε, κάποια όρια για την ε, οικογενειακή επανένωση, κάποια ε, κάποιες ε, προδιαγραφές οι οποίες θέλουν να αποτρέψουν τους ε, γάμους δια της βίας, τους υποχρεωτικούς γάμους. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν ανησυχίες σε ορισμένα κράτη-μέλη. Αν κατάλαβα λοιπόν καλά, αναφερθήκατε ότι υπάρχει αυτή η εταιρική σχέση για την κινητικότητα ώστε να, στα πλαίσια της καλύτερης πρόσβασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση που πρέπει να υπάρξει. Πέραν λοιπόν την, της εφαρμογής των συμφωνιών για την εκπαίδευση και των δυνατοτήτων εργασίας υπάρχουν και κάποια κοινωνικά θέματα τα οποία πρέπει να ρυθμιστούν και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Στην ε, δική μου χώρα, στη Γερμανία, αντιμετωπίζουμε μεγάλη αγανάκτηση της ε, κοινή γνώμης εξέγερση της κοινή γνώμη ουσιαστικά, διότι υπάρχει η εντύπωση ότι είναι υπερφορτωμένο το κοινωνικό σύστημα προνοίας και ιδίως των Δήμων και κοινοτήτων λόγω της ζωής πολιτών της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Αν λοιπόν υπάρξει αυτή η συμφωνία κινητικότητος και υπάρξει πρόσβαση των ανθρώπων που έρχονται στη Γερμανία και στις κοινωνικές πρόνοιες, τότε ουσιαστικά θα μας πλημμυρίσουν αυτοί οι άνθρωποι και θα μείνουμε χωρίς δυνατότητες υποδοχής. Γι' αυτό θα ήθελα να θέσω το ερώτημα πώς αντιμετωπίζει το Συμβούλιο, ποιες είναι οι θέσεις στο Συμβούλιο για τα θέματα φιλελευθερωποίησης προξενικών θεωρήσεων. Θα ήθελα κάτι συγκεκριμένο να μου πείτε. Ευχαριστώ κύριε Ζόμερ. Τελειώσαμε τον κατάλογο των συναδέλφων που ήθελαν να μιλήσουν. Μου είπαν ότι δεν θέλει να πάρει το λόγο το Συμβούλιο. Υπάρχει κάποιος παρόν εκπρόσωπος του Συμβουλίου που θέλει να προβεί σε κάποια σχόλια έχοντας ακούσει τη συζήτηση. Όχι. Κύριε Μαντσοβίζη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Ε, Όσον αφορά το Μαρόκο, το ρώτησε η κυρία Ζόμερ. Ελπίζω ότι να μην υπάρχει ένα απομένον πρόβλημα με το Μαρόκο. Το τελευταίο σημείο στη συζήτηση ακριβώς αφορούσε κάποιες ανησυχίες περί δυνατότητας μεταφοράς κοινωνικών δικαιωμάτων και η δυνατότητα του Μαρόκο να μπορεί να έχει την προπτική να μην χρειάζονται οι υπήκοοι του, οι του θεωρήσεις. Το βασικό, μάλλον έχουμε δύο, βασικά στοιχεία. Πρώτα απ' όλα έχουμε την επανεισδοχή, τη συμφωνία επανεισδοχής, εδώ και χρόνια είχε κολλήσει αυτή και έχει γίνει πλήρως αποδεκτή σαν στόχο και θέμα διαπραγματεύσεων και για επικόστη των χωρών. Και θα ήθελα να πω και το άλλο. Το να υπάρχουν σαφείς στόχοι στην εταιρική σχέση είναι απαραίτητο για να προστατεύονται αυτοί που για κάποιο λόγο έχουν κολλήσει στο Μαρόκο, έχουν απομονωθεί στο Μαρόκο. Θέλω να αναφέρεται η σύμβαση της Γενέβης και όλοι οι κανόνες που αφορούν τη διεθνή προστασία δεν διαπραγματευόμεθα με το Μαρόκο νομικές υποχρεώσεις αλλά στόχους και γι' αυτό είναι σημαντικό το, το θέμα αυτό. Διευκόλυνση χορηγήσεως προξενικών θεωρήσεων ενδεχομένως επανεισδοχή. Είναι ανοιχτή συζήτηση. Η αντιμετώπιση εκείνων που είναι πρόσφυγες ή παράνομοι στο Μαρόκο και προφανώς παραμένουν σε μια κατάσταση ε, που μπορεί ανοιχτά να επικρίνεται. Αυτό είναι ένα θέμα που συζητείται και έχει γίνει αντιληπτό από τους εταίρους μας. Νομίζω ότι από αυτής της βάσης μπορώ να είμαι αρκετά αισιοδόξο. Θα μπορεί να μην έχουμε, μάλλον δεν θα έχουμε άλλα προβλήματα. Πιο συγκεκριμένα μπορώ να σας πω στην επόμενη εβδομάδα, την επόμενη εβδομάδα όταν θα ολοκληρωθούν οι συζητήσεις. Αυτή είναι η κατάσταση μέχρι τώρα και αυτό είναι αρκετά σημαντικό. Μιλισμονούμε ότι όταν μιλάμε για νόμιμη μετανάστευση, μεταφορά δικαιωμάτων, αναγνώριση, όλα αυτά ε, καλύπτονται από δράσει σε διμερέ επίπεδο με τα κράτη-μέλη. Εμεί δεν έχουμε αρμοδιότητα σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά άδεια εργασία, συνθήκε εργασία. Έχουμε αρμοδιότητα όσον αφορά ε, παραμονή, διαμονή κλπ. Όλα αυτά γίνονται διμερώ με τα κράτη-μέλη, εξού και σημασία να έχουμε πολλά κράτη-μέλη που συμμετέχουν. Διαφορετικά δεν μπορούν να ολοκληρωθούν τα δύο αυτά προγράμματα. Όσον αφορά την Τουρκία, το αναφέρατε νομίζω. Το, της χαλαρής πολιτικής όσον αφορά τις θεωρήσεις που ακολουθεί η Τουρκία. Μπορεί να μπει κανείς στην Τουρκία και χωρίς θεωρήσεις σε πολλές περιπτώσεις. με πολύ χαμηλό τίμημα από πολλές χώρες που μπορούν να μπουν χωρίς θεώρηση. Αυτό θα συμπεριληφθεί σε μελλοντικό διάλογο για την ε, διευκόλυνση χορηγήσεως ε, θεωρήσεων. Λέμε ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να εξεταστεί λόγω της πολιτικής αυτής για τις θεωρήσεις που συμβάλλει στο να παράγει πάρα πολλούς παρανόμους μετανάστες που βρίσκονται στην ε, Ελλάδα. Εδώ δεν μπορούμε να επιβάλλουμε το κεκτημένο Μπορούμε να το συζητήσουμε όμως, να δούμε πώς θα πετύχουμε το ευκταίο αποτέλεσμα. Να μην συμβαίνει αυτό το φαινόμενο. Και είναι πρόθυμες οι τουρκικές αρχές να το συζητήσουν. Θα δούμε από τη στιγμή που θα ξεκινήσουν οι συνομιλίες τι θα γίνει. Αλλά είναι, συμπεριλαμβάνεται αυτό το θέμα συνομιλίες. Τώρα αν καταλαβαίνω σωστά, μετά αναφερθήκατε στα όσα συμβαίνουν εντός της Ενώσεως, κυρίως στην Ελλάδα και σε άλλες νότιες χώρες που φιλοξενούν ούτω υπήν ε, του ετούντε άσυλο και του πρόσφυγε. Έχουμε ευρωπαϊκό, ευρωπαϊκή νομοθεσία, επιβάλλεται. Έχουμε ξεκινήσει κάποιε δικασίε κατά παράβαση κατά κάποιων χωρών, κυρίω όσον αφορά τι συνθήκε φιλοξενία. Παρακολουθούμε μετά άμεσα και με την ΕΑΣΟ στο, άρθρο 333 του νέου κανονισμού του Δουβλίνου αναφέρεται το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης με σχέδιο δράσης που πρέπει να εφαρμόζεται κλπ. κλπ και χρησιμοποιούμε και τα διαθέσιμα χρήσιμα για να υποστηρίξουμε σχετικές προσπάθειες. Στην Ελλάδα, παραδείγματο χάρη, υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο δράσης με συγκεκριμένα αποτελέσματα ορατά. Η κατάσταση παραμένει δυσχερέστατη. Το ξέρω. Δεν θέλω να πω ότι έληξε το πρόβλημα. Αντιθέτω, πόρα απέχει από αυτό. Αλλά η διαδικασία τουλάχιστον έχει ξεκινήσει. Αναφέρω στο, ε, αναμένω εντάσει στο μέλλον, διότι εκτίθενται περισσότερο οι νότιε χώρε. Οπότε θα πρέπει να δείξουμε μεγαλύτερη αλληλεγγύη προς αυτές τις χώρες. Διότι κρατάνε τα σύνορα εκ μέρους ε, της υπόλοιπης Ένωσης. Και το νέο οικονομικό μέσο προτείνουμε αυτή τη φιλοσοφία ακολουθεί. Να αντιμετωπιστούν οι χώρες, ε, να είναι προστάτες των συνόρων της Ένωσης αυτές οι χώρες. Αυτό κάνουμε. Λοιπόν, υπάρχουν κάποια αποτελέσματα, αλλά συμφωνώ, ακόμα απέχουμε από τη βέλτιστη κατάσταση. Η ΆΣΟ έχει λίγα, λίγους πόρους, αλλά δεν μπορεί να περιμένει κανείς ένα μικρό φορέα να αναλάβει όλο αυτό το σύστημα. Δεν δημιουργήθηκε γι' αυτό, δημιουργήθηκε για να βοηθήσει κινητοποιώντας δυναμικό στα κράτη-μέλη, ούτως ώστε να αντιμετωπίζονται κρίσιμες καταστάσεις. Δεν είναι υπηρεσία για διαθωτικές παρεμβάσεις. Εν πάση περιπτώσει, συνεχώς καταβάλουμε προσπάθειες με αυτό το φορέα για να βελτιώσουμε και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, που τώρα ξεκίνησε για το θέμα της επανεισδοχής στη Νότια Οσετία, να Γκόρνο Καραμπάχ κλπ. Η συμφωνία επανεισδοχής εξαρτάται επί απλής αρχής και απλών κανόνων. Πρώτα απ' όλα θέμα υπηκότητας που θα πρέπει να διαπιστώνεται μέσω εγγράφων ή μέσω άλλων μέσων θα πρέπει να διαπιστώνεται, να εξακριβώνεται. Μιλάμε για Οριανούς, Αρμενίους πολίτες που διαπιστώνεται ότι έχουν αυτή την υπηκότητα. Δεύτερον, πολύ σημαντικό, εάν η επανεισδοχή δεν ε, υπονομεύει τα δικαιώματά τους, τα θεμελιώδη δικαιώματά τους. Δεν είναι μια αυτόματη διαδικασία, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και ποια είναι η κατάσταση που θα επικρατήσει όταν επιστρέψουν στη χώρα και κάποιοι από αυτοί ζητάνε και άσυλο. Δεν έχω στοιχεία όσον αφορά το ποσοστό αποδοχής των αιτήσεων ασύλου από Αρμενία και Γεωργία, αλλά ε, έχουν, ε, γίνονται αιτήσει, άρα δεν είναι αυτόματη η επανεισδοχή, δηλαδή τους επιστρέφουμε σε δύσκολες περιοχές και περιφέρειες. Οι περιφέρειες, οι περιοχές δεν έχουν τόσο μεγάλη σημασία. Ε, έχουμε συμφωνίες με μια χώρα για υπήκο της χώρας. Τώρα για το Πακιστάν. Να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Η συμφωνία της Ένωσης με το Πακιστάν μέχρι τώρα έχει δώσει ελάχιστα αποτελέσματα, το είπα στην αρχή και το επαναλαμβάνω τώρα. Γιατί πιέζω τις πακιστανικές αρχές να, να έρθουν στην Επιτροπή, τη Μιχτή Επιτροπή για την επανεισδοχή, γιατί πρέπει να καθορίσουμε κάποιους όρους. Διότι τώρα αυτοί που επιστρέφουν ε, εντάσσονται μέσα σε διμερείς συμφωνίες κάθε χώρας με το Πακιστάν. Το πρόγραμμα που αναφέρατε θα υλοποιηθεί τους επόμενες, ε, ε, ε επόμενους μήνες και χρόνια, μεταξύ άλλων από την ΥΠΑΤΗ Αρμοστία για τους πρόσφυγες και είναι κάτι που γραμμίζουμε και στην έκτη αξιολόγηση. Πρέπει να προσέξουμε περισσότερο τι γίνεται σε εκείνους που επιστρέφουν στη χώρα τους. Τι συμβαίνει μετά όταν επιστρέψουν. Αυτό το πρόγραμμα έχει στόχο αυτό. Να αντιμετωπιστεί η πιο δύσκολη περίσταση. Αυτή του Πακιστάν ακριβώς. Ίσως έτσι θα μάθουμε και για άλλε χώρε τι μπορούμε να κάνουμε. Στα πλαίσια του ΕΑΖΟ, όταν συζητάμε τη τι εκθέσει χώρα καταγωγή όπω αποκαλούνται, ασχολούμεθα και με αυτό. Δηλαδή να εντοπίσουμε ακριβώ ποια κατάσταση αντιμετωπίζουν αυτοί οι άνθρωποι όταν πιστεύονται σε χώρε που πιθανότατα οι χώρε αυτέ οι ίδιε θέλουν ετούντε άσυλο. Και κάποιοι αυτοί που υποβάλλουν τα έτοιμα άσυλο απορρίπτονται, του επιστρέφουμε και μετά πρέπει να επανενταχθούν στην κοινωνία τη χώρα του. Αυτό το κοιτάμε, το ελέγχουμε. Δεν λέω ότι είναι τέλεια η κατάσταση, έχουμε επίγνωση Διαθέτουμε προσπάθεια, πολιτική βούληση και μέσα για να κάνουμε περισσότερα. Το ίδιο ισχύει και για, τους, για τη ρήτρα για του υπηκόου των χωρών. Είπαμε στην έκθεση αξιολόγηση κάνα δύο πράγματα. Πέρα αυτού που είπα τώρα. Πρώτα απ' όλα, δεν θέλουμε μεμονωμένε συμφωνίε επανεισδοχή χωρί κάποια διευκόλυνση. Αυτό κάνουμε τώρα. Διότι δεν πιστεύουμε ότι απλώ είναι δίκαιο να μιλάμε απλώ για επανεισδοχή, ούτε δίνει και κάποια κίνητρα. Μετά, είπαμε υπήκος τρίτης χώρας όταν αυτό ενδείκνυται για τους υπηκός τρίτων χωρών. Και δεν προτείναμε να επιστρέψουμε υπηκός τρίτων χωρών στην Αρμενία, στη συμφωνία με την Αρμενία, αλλά δεν μας υποστήριξε το Συμβούλιο. Υποχρεωθήκαμε να ακολουθήσουμε την εντολή που αφορά και την επανεισδοχή για υπηκός τρίτων χωρών. Ακόμα και με μια χώρα που δεν, με μια χώρα που δεν έχει κοινά σύνορα. Ξέρετε ποια είναι η διαδικασία χορηγήσεως εντολής. Δόθηκε συγκεκριμένη εντολή να καλύπτονται και οι υπήκοοι χωρών και εφαρμόζουμε την εντολή που μας δόθηκε. Όσον αφορά την Τουρκία, να τα πούμε με το όνομά τους τα πράγματα. Οι τουρκικές αρχές ξέρουν ότι θα ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις και το διάλογο για το ενδεχόμενο αποτέλεσμα που, ακολ, αποκαλείται απελευθέρωση από τη χορήγηση θεωρήσεων φιλελευθεροποίηση της θεωρήσεων από τη στιγμή που θα συναυθεί και συμφωνία επανεισδοχής. Πρώτα, αυτοί όταν θέλουν να τα αντιστρέψουν ε, πρέπει να το καταλάβουν ότι δεν γίνεται. Πρέπει να είναι συμμετρική ε, η προσέγγιση, να υπάρχει συμφωνία επανεισδοχής μαζί και μετά να απελευθερωθεί αυτή η ανάγκη ε, για να μειωθεί η απέτηση για τη χορήγηση βίζας. Λοιπόν, για τους υπηκόστητων των χωρών το είχαμε κάνει αυτό με την Ρωσία, την Ουκρανία κλπ. Πολύ συχνά υπάρχει κάποιο κενό μεταξύ της θέσης ισχύ της επανεισδοχής για τον υπήκο της χώρας και τη θέση σε ισχύ της ρήτας που καλύπτει τους υπηκόστητων των χωρών. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Μετά, πάντα υπάρχει ένα αντάλλαγμα. Για όλους τους κανόνες για διευκόλυνση, φιλελευθεροποίηση, συμφωνία διευκόλυνση θεώρηση, δηλαδή να μπορεί να ταξιδέψουν αυτοί και χωρίς θεώρηση, προηγείται αυτή πλήρη αξιολόγηση τη συμφωνία επανιστοχή που θα πρέπει να εφαρμόζεται πλήρω. τεχνικός πώ δεν θα μπορούσε να αρθεί η απέτηση θεώρηση με την Τουρκία αν πριν δεν έχει εφαρμόσει πλήρω η Τουρκία όλε τη συμφωνία για πανεισδοχή συμπεριλαμβανομένη και τη ρήτρα που καλύπτει η πικόστη των χωρών. Αυτή η ασυμμετρία υπάρχει τώρα και θα εξακολουθήσει μετά εκτό και εκτό, το υπογραμμίζω, εκτό. Το ότι ξεκινά διάλογο δεν σημαίνει ότι θα μειωθεί η χρονική διάρκεια που απαιτείται. Ας μην πιέζουμε τις καταστάσεις όμως. Πρέπει να δημιουργηθεί κλίμα εμπιστοσύνης στις συνομιλίες πρώτα. Αλλά πιστεύω ότι όταν συζητήσουμε για την άρση απαιτήσεως για θεώρηση, τότε πιστεύω ότι θα τεθεί, όχι σίγουρα, θα τεθεί και το θέμα της επανεισδοχής υπηκότητων των χωρών. Θα ήταν δίκιο να συζητηθεί, διότι αυτούς κανόνες ακολουθούμε. Ότι θα απελευθερώσουμε τις θεωρήσεις από τη στιγμή που θα εφαρμόζονται πλήρως οι συμφωνίε επανεισδοχής. Άρα ε, υπάρχει μια κάποια ισορροπία. Έχουμε κάποιες πληροφορίες για τα τεκτενόμενα εντός Τουρκίας. Η Τουρκία λειτουργεί αρκετά καλά. Χρησιμοποιεί και σωστά και τα χρήματα που της δίνουμε στα πλαίσια του ε, προενταξιακού μέσου ε, για να διευκολύνουμε εκείνους που είναι παράνομοι και τους σταματάνε έχουν χτίσει εγκαταστάσει με χρήμα τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω, χώρου υποδοχή όπου φιλοξενούνται οι άνθρωποι οι οποίοι συλλαμβάνονται στα σύνορα, μπαίνουν παράνομα. Και που φιλοξενούνται και οι πρόσφυγε. Μπορεί όμω και οι πρόσφυγε να γίνουν και στο μέλλον και μια απειλή, να γίνουν παράνομοι μετανάστε που θέλουν να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα το συζητήσουμε του Τούρκου. Και οι Τούρκοι το αναγνωρίζουν αυτό. Και από τη στιγμή που θα ξεκινήσει ο διάλογος θα δούμε και πώς θα πετύχουμε το στόχο. Όσον αφορά την επιβολή του νόμου και όσον αφορά τη φιλοξενία των προσφύγων κάνουν ποιοτική δουλειά. Όσο το συζητάμε ανεπίσημα είναι δύσκολο να δούμε και τι γίνεται. Τη στιγμή θα καθίσουμε και θα συζητήσουμε το θέμα επίσημα για να πιστούμε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για να απελευθερώσουμε την απέτηση για θεωρήσεις τότε μπορούμε να προσμετρήσουμε τα αποτελέσματα λεπτομερέστερα. Τώρα, όσον αφορά την κατάσταση στο Συμβούλιο με την Τουρκία. Η κατάσταση στο Συμβούλιο είναι σαφής. Η Τουρκία έχει, ε, έχει ευλογηθεί ο δικός χάρτης για απελευθέρωση της θεώρησης με την Τουρκία. Εδώ και μήνε. Από τη στιγμή που η Τουρκία θα υπογράψει και θα εφαρμόσει τη συμφωνία επανεισδοχή. Αυτό κάνουμε τώρα, ώστε να καταλήξουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Υπάρχει ένας φόβος από την τουρκική πλευρά. Λένε εντάξει είναι η αρχή μιας διαδικασίας. Πότε είναι το τέρμα της διαδικασίας. Τα κράτη-μέλη τότε θα είναι έτοιμα να εθετήσουν μια πρόταση που θα είναι να αλλάξει το καθεστώς της Τουρκίας. Δεν υπάρχει εγγύηση. Θα θυμόσαστε ότι είναι μια απόφαση που ελήφθη από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με ειδική πλειοψηφία. Και η καλύτερη εγγύηση είναι ότι Εάν γίνει ένας διάλογος με βάση στοιχεία και αποδειχθεί ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για να υπάρχει εμπιστοσύνη, εμείς θα κάνουμε πρόταση. Και αν κάνουμε πρόταση, εννοείται ότι θα την υπερασπιστούμε, διότι θα είμαστε πεπισμένοι ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις. Τότε θα ακολουθηθούν και οι διάφοροι διοργανικοί κανόνες. Αυτή είναι η μόνη εγγύηση για δικαιοσύνη που μπορούμε να δώσουμε. Και αυτό το βλέπει η Τουρκία, το καταλαβαίνει η Τουρκία. Δεν ξέρω αν ξέχασα κάτι. Φαντάζομαι ότι όλες οι ερωτήσεις έχουν απαντηθεί και ως εκ τούτου μπορώ να κλείσω τη συζήτησή μας. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ματσερίτσι. Ερχόμαστε στο επόμενο σημείο της ημέρας της διάταξης. Έχουμε μια μικρή προπορία χρονική και θα ήθελα να προτείνω δεν ξέρω πώς νιώθετε εσείς αλλά δεν είναι η κατάλληλη θερμοκρασία για μια συνεδρίαση παθαίνουν πνευμονία ορισμένοι βήχουν Είναι πολύ ζεστά εδώ. Αυτό δείχνει την πολυμορφία της αντίληψης της, θερμο, της θερμοκρασίας. Από ό,τι ξέρω πάντως η κυρία Ματιού είναι έτοιμη να κάνει την παρουσίαση του θέματος του κυρίου Λούχαν το σημείο 38. Καταρχήν, συγγνώμη, να σας πω ότι η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών στο σχέδιο εκθέσεως του κυρίου Μαρινέσκου για την διευκόλυνση προξενικών θεωρήσεων με την Μολδαβία είναι στις 8, 28 Φεβρουαρίου 6 ώρα το απόγευμα. Την επόμενη Πέμπτη στις 6 το απόγευμα. Αν συμφωνείτε λοιπόν με, το, με την πρότασή μου, συνεχίζουμε με την ημερήσια διάταξη και θα ήθελα να ζητήσω από την κυρία Ματσιού να παρουσιάσει το θέμα του κυρίου Λούχαν για τα έγγραφα που αφορούν τα επενδυτικά προϊόντα. Μπορούν οι κυρίες στο πίσω μέρος της να σιωπήσουν ενδεχομένως. Κέρια έγγραφα με βασικές πληροφορίες σε σχέση με επενδυτικά προϊόντα επί τη βάση του εγγράφου της Κομισιόν του Ιουλίου του 2012 για ένα κανονισμό για τα, τις βασικές πληροφορίες σε σχέση με τα επενδυτικά προϊόντα. Ο στόχος αυτής της πρότασης είναι η βελτίωση της διαφάνειας και η διευκόλυνση της συγκρισιμότητας μεταξύ των χρηματοπιστωτικών προϊόντων για τους επενδυτές. Δεν, α, η Επιτροπή Οικονομικών Θεμάτων είναι η αρμόδια επί της αρχής και η συγγήτρια είναι η κυρία Μπέρες. Κυρία Ματιέ, σας δίνω το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη για τον κύριο Λούαν, ο οποίος χρειάστηκε να φύγει να πάει στη Ρουμανία. Και έχει προετοιμάσει ένα κείμενο το οποίο θα διαβάσω. Οι λιανικού χαρακτήρα επενδυτές που θέλουν να κάνουν μια επένδυση έχουν όλο και περισσότερα προϊόντα από τα οποία να επιλέξουν. Πολλές φορές τα προϊόντα αυτά προτείνουν συγκεκριμένες διαδικασίες επενδυτών που είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες των επενδυτών αλλά είναι δυσνόητες πολλές φορές. Παρακαλώ όλους αυτούς που θέλουν να ανοίξουν πηγαδάκι να πάνε έξω από την Οι πληροφορίε λοιπόν οι οποίε πρέπει να δοθούν αυτή τη στιγμή στου ε, επενδυτέ σε σχέση με τα προϊόντα δεν είναι αντικείμενο συντονισμού και πολλέ φορέ δεν βοηθούν τη σύγκριση διαφορετικών προϊόντων και την α, κατανόηση των χαρακτηριστικών του. Πολλέ φορέ οι επενδυτέ, οι μικροεπενδυτές κάνουν επενδύσει χωρί να καταλαβαίνουν το χαρακτήρα αυτών των επενδύσεων και υφίστανται απώλειες ως εκ τούτου. Οι διατάξεις για την διαφάνεια των προϊόντων που προσφέρονται σε μικροεπενδυτέ είναι ένα σημαντικό μέτρο προστασία και αυτό είναι μια απαράγραπτη προπόθεση για να μπορέσει να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών. Η πρόταση του κυρίου Λουάν τονίζει τα θεμελιώδη δικαιώματα τα οποία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να τη χάνουν σεβασμού. Προτείνει ο κ. Λούαν τα κράτη-μέλη να αναλάβουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν ότι υπάρχουν διοικητικού χαρακτήρα οι οποίες θα δημοσιεύονται μόνο όταν αυτό είναι απαραίτητο και να διαγράφονται όταν εκπνεύσουν. Το να έχουμε κυρώσεις οι οποίες διακούν πολύ χρονικό διάστημα μπορούν να οδηγήσουν σε αρνητικά αποτελέσματα και να στιγματίσουν ένα άτομο χωρίς να λάβουν υπόψη την προηγούμενη του συμπεριφορά. Ευχαριστώ πολύ. <clears throat> Δεν βλέπω εδώ η Κομισιόν ή το Συμβούλιο να θέλουν να λάβουν το λόγο. Όχι. Κάποιος από τους συναδέλφους θα ήθελε να λάβει το λόγο. Κύριος Χούτερ. Εγώ χαιρετίζω την πρόταση αυτή της Κομισιόν. Ένα τμήμα της ε, χρηματοπιστωτικής ε, κρίσης είναι ότι υπήρξαν πολλά προϊόντα που αγοράστηκαν χρηματοπιστωτικά από τους πολίτες που δεν θα έπρεπε να τα είχαν αγοράσει. Επομένως είναι ε, καλό δεχτεί αυτή η πρόταση γιατί βοηθάει και αυτούς οι οποίοι χρειάζονται <clears throat> νομική αρρωγή γιατί αναστρέφει το βάρος απόδειξη ότι πρέπει αυτός ο οποίος παρέχει τα ε, επενδυτικά προϊόντα να εξηγήσει περί τίνος πρόκειται και να αποδείξει ότι δεν έχει παραπλανήσει. Βλέπω όμως ότι η Κομισιόν κάνει πολλές εξαιρέσεις στα σημεία 2α, β, και δ εμείς θεωρούμε ότι αυτές οι εξαιρέσεις θα πρέπει να διαγραφούν και για τη δημοσίευση των κυρώσεων θα πρέπει να είναι σαφές ότι πρέπει να δια... δημοσιευθούν αυτές οι κυρώσεις ώστε να εξασφαλιστεί η απαραίτητη διαφάνεια και αυτό σε περιπτώσεις που ε, μπορούν να διακινδυνεύσουν βέβαια την ε, ασφάλεια της αγοράς θα πρέπει να διαγράφονται όταν περάσει η περίοδος εφαρμογής τους. Και επίσης θα πρέπει όλα αυτά να υπόκεινται στην προστασία της οδηγίας για τα προσωπικά δεδομένα. Και κάτι ακόμα το οποίο είναι σημαντικό για μένα είναι να μπορέσουμε να έχουμε τις ομάδες στόχου για τις οποίες θα πρέπει να παρέχεται ε, τυποποιημένη πληροφόρηση. η προηγούμενη οδηγία MIFID καθορίζει αυτές τις ομάδες στόχου και θα πρέπει να υπάρχει και κάποια επεξήγηση γιατί ένα προϊόν ε, προσαρμόζεται προς τις ανάγκες μιας ομάδος επενδυτών. Και φυσικά ένα από τους βασικούς στόχου που θα πρέπει να εξυπηρετούμε πάντα θα είναι η προσπάθεια να μειώνεται η πολυπλοκότητα των χρηματοπιστωτικών προϊόντων και να γίνονται πιο εύκολα αναγνώσιμα και κατανοήσιμα. Από τους επενδυτέ. ναι, σας ευχαριστώ λέει πρόεδρο. Κάποιο άλλο θέλει να λάβει το λόγο, όχι. Προθεσμία για τις τροπολογίες 27 Φεβρουαρίου ή δεν υπάρχει κάποια προθεσμία. Θα ληφθεί η απόφαση την επόμενη εβδομάδα. Εντάξει, θα σας ε, κοινοποιηθούν όλα αυτά. 27 Μαρτίου, κατά πάσα πιθανότητα. 20-21 Μαρτίου θα γίνει ψηφοφορία. Ερχόμαστε τώρα σε ένα σημείο της τη διάταξης που είναι και κλεισμένο το θυρών. Η κυρία Λεμπέη δεν είναι παρούσα, είναι στο δρόμο. Σας ζητώ λοιπόν να διακόψουμε για πέντε λεπτά με την ελπίδα να μπορέσει να έρθει και να αντιμετωπίσουμε αυτό το τελευταίο σημείο στην μέση διάταξη. Πέντε λεπτά διακόψουμε. Um, Καταφτάνει η κυρία Λεμπάη. Οπότε we Οπότε συνεχίσουμε και σας ασχοληθούμε το σημείο, σημείο, τελευταίο σημείο της, Αμερι... της Διάταξης και κλεισμένο των θυρών. Παρακαλώ όλους όσους δεν έχουν το δικαίωμα να είναι παρόντες κατά τη διάρκεια συνεδριάσου και κλεισμένο των θυρών να αποχωρήσουν παρακαλώ από την αίθουσα.